τα προϊόντα καπνού. Θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Γεωργίευα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την πρόσκληση να καταθέσουμε μια δήλωση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι συμφωνίε για την εμπορία προϊόντων καπνού. Οι συμφωνίε αυτέ με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου σε ένα μέσο και εργαλείο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Η πρώτη υπεγράφει το 2004. Έκτοτε και μέχρι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο βασικός μας σύμμαχος στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων που είναι ε, μια εγκληματική πράξη αξιόπινη ε, που στερεί πάρα πολλά έσοδα από τους προϋπολογισμούς μας. Έχουμε τα στοιχεία γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο διαφυγόντα κέρδη και έσοδα για το κράτη κυρίω λόγω του λαθρεμπορίου. Αλλά δεν είναι μόνο ο προϋπολογισμός των κρατών μελών, είναι και τη Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττεται. Για να το δούμε λοιπόν σε ένα πλαίσιο, τα 28 κράτη-μέλη το 2013 είχαν φορολογικά έσοδα από νόμιμες πωλήσει καπνού πάνω από 90 δις ευρώ. Σημαίνει ότι έχουν χάσει πάνω από 10% του εισοδήματος που θα ήταν υπέρ των πολιτών λόγω αυτής της παρανομίας και της δραστηριότητας λαθρεμπορίου. Άρα η κατεπολέμηση ε, του λαθρεμπορίου τσιγάρων έχει και πολύ σημαντικό ε, οικονομικό ε, στόχο. Επίσης ξέρουμε και τι σημαίνει για τη δημόσια υγεία η εθνική νομοθετική περιορισμοί και οι υψηλέ τιμέ έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν του πολίτε από το κάπνισμα και να προστατεύουν ιδίω του νέου. Σε αντίθεση με αυτά, τα παράνομα τσιγάρα διατίθενται και για τους νέους ε, και είναι σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Υπάρχει και ένα στοιχείο, μια διάσταση ασφαλείας, αφού το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι από τις βασικές πηγές εισοδήματος για το οργανωμένο έγκλημα. Και όπως γνωρίζετε, στις 28 Απριλίου εγκρίναμε μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα, ένα θεματολόγιο ασφαλείας, προσπαθώντας να περιορίσουμε το εισόδημα από παράνομες δραστηριότητε σε διάφορες ομάδες και μεταξύ αυτών είναι και το λατρεμπόριο προϊόντων καπνού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει πλήρως ε, την ανάδειξη αυτής της ε, καταπολέμησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Για ποιο λόγο, διότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και απαιτεί μια παγκόσμια λύση. Αυτό που έχουμε τώρα ένα πρωτόκολλο στη Συμφωνία Σύμβαση του ΠΟΕ για τον έλεγχο και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας πω ότι στις 4 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση προς το Συμβούλιο να κυρώσει αυτή τη σύμβαση και το πρωτόκολλο. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί χρόνο αυτή η κύρωση. Και μέχρι τώρα χρειάζονται 40 ε, κράτη να ε, το κυρώσουν για να τεθεί σε ισχύ και μόλις 7 έχουν εγκρίνει. Και ακόμα και αν φτάσουμε στα 40 κράτη-μέλη για να τεθεί σε ισχύ αυτή η σύμβαση, δεν γνωρίζουμε ακόμα εάν οι βασικές χώρες που είναι χώρες προέλευσης και διέλευσης διαμετακόμισης θα υπογράψουν. Σας διαβεβαιώ ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά το ρόλο μας για να ενθαρρύνουμε, να παροτρύνουμε ακριβώς αυτές τις χώρες να κυρώσουν εν γέρος το λόγο πρωτόκολλο. Επίσης προχωρούμε έγκαιρα ε, στην εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Ωστόσο η οδηγία αυτή δεν μπορεί να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο της ε, στο λαθρεμπόριο τσιγάρων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυτή τη χρονική στιγμή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε σχέση με αυτό που εμείς θα επιδιώκαμε και θα αποσκοπούσαμε ως πιο μακροπρόθεσμο στόχο. Και Έχουμε και άλλα μέσα στη ε, διάθεσή μας ε, που είναι συμφωνίες με τις μεγάλες ε, εταιρείες καπνού. Το 2004 υπογράψαμε με τη Philip Morris International. Εκπνέει η συμφωνία αυτή τον Ιούλιο του 2016 και εισήγαγε καινοτόμα μέσα τη δέουσα επιμέλεια, το να ξέρεις ποιοι είναι οι αγοραστές, οι πελάτες σου και να είναι και προσβάσιμη η δημόσια αυτή η πληροφορία και κάποια άλλα στοιχεία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Φίλιπ Μόρις συμφώνησε να πληρώσει 1,25 δισεκατομμύρια και 90,3% ε, αυτού του ποσού ε, πήγε προς τα κράτη-μέλη. Η συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική και μπορεί να συμπεριλάβει και κάποια άλλα στοιχεία που δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εύκολα με νομοθετική οδό. Ιδιαίτερα ε, να ε, πληρώνουν πρόστιμα σε περίπτωση κατασχέσεων ε, για να συμμορφωθούν. Και είναι ένα κίνητρο αυτό. Ο κύριος Σεμετά, προκάτοχός μου, ήδη έχει ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι είχαμε με τη Philip Morris International σύντομες διερευνητικές επαφές όπου η εταιρεία ε, θέλησε να συζητήσει, δήλωσε προθυμία, εν να συζητήσει παράταση της συμφωνίας. Και ξέρουμε τώρα ότι η μεγαλύτερη μάστιγα δεν είναι αυτές οι εταιρείες, αλλά είναι ε, τα φτηνά ε, τσιγάρα που πουλούνται στη Λιανική, στο όλα Στη συνέχεια λοιπόν, ανάλογα με τις εξελίξεις και τη στάση των εταιριών, θα δούμε τι μέλλον θα έχουν αυτές οι συμφωνίες. Θα ολοκληρώσουμε μια, την αξιολόγηση σε λίγες εβδομάδες, την οποία βεβαίως θα υποβάλουμε και στο Κοινοβούλιο, αλλά και θα τη δημοσιεύσουμε. Υπάρχουν στοιχεία ξεκάθαρα ότι βασικός στόχος της συμφωνίας με τη Φίλιπ Μόρις, που είναι η μείωση ε, των λαθρέων τσιγάρων Φίλιπ Μόρις στη μαύρη αγορά έχει επιτευχθεί από το 2006 μέχρι το 2014 ο όγκος των παρανόμων των πλαστών λαθρέων τσιγάρων PMI έχει ε, πέσει κατά 85% και αυτό ε, ξεπερνάει κατά πολύ το μέσο όρο των κατασχέσεων. Αυτό αφορά το λαθρεμπόριο των τσιγάρων Φίλιπ Μόρις που μπορεί να είναι και γνήσια προϊόντα αλλά και πλαστά. Ε, σκεφτόμαστε πώς θα προχωρήσουμε τώρα, εξετάζουμε τα επόμενα βήματά μας με γνώμονα την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολιτών μας. Ε, είναι ανοιχτή έκβαση, ε, είμαστε πρόθυμοι και εμείς και ανοιχτοί και να συζητήσουμε και είναι πολύ σημαντικά τα όσα θα ακούσουμε σήμερα από εσά για να συνεισφέρετε στις διαβουλεύσεις και στις συζητήσεις μας θα σας ε, τηρώ απολύτως ενήμερους όσο προχωρά αυτή η διαδικασία για το τόσο σημαντικό ζήτημα όσο και ευαίσθητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή βλέπω ότι παρευρίσκεται... How do I pronounce Ο κύριος Γκάιερ, θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ του πρασίνους για την πρωτοβουλία. Αλλά ο κύριο Γκάιερ είναι στη σοσιαλιστική ομάδα. Δεν είστε μέλο των πρασίνων. Όχι. Πού είναι η πράσινη τότε. Hey, I got, I'm sorry, I got confused, I apologize. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Δεν έπρεπε να το πω. Έπρεπε να σταματήσω όταν ήταν η ώρα να σταματήσω. Ε, Παραμίλησα. Ευχαριστώ πολύ. Well, we'll sort it out anyway later. Εντάξει, το λύσαμε το θέμα. Ευχαριστούμε την κυρία Γεωργίευα. Ο κύριος Σάρβαμα, για δύο λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω, προφανώς, για αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Το εκτιμούμε. Εκτιμούμε ότι ήρθατε στο Κοινοβούλιο με μία δήλωση για τη συνεργασία και τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεγάλες εταιρείες ε, καπνού και παραγωγής τσιγάρων. Κατά την απόψή μας, διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κομισιόν και των εταιρεών αυτών θα, είναι, θα έπρεπε να είναι ε, πολύ πιο ανοιχτές και πολύ πιο διαφανείς. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μας επετράπει να δούμε τα έγγραφα μέσα σε ένα δωμάτιο μόνο καμιά, για καμιά δύο ώρες. Και αυτό έγινε μετά από ανταλλαγή επιστολών με τον προκάτοχό σας. Όμω χρειάζεται εξειδικευμένο δικηγόρο για να καταλάβει οτιδήποτε έχουν, έχει γραφτεί σε αυτά τα έγγραφα. Τώρα περιμένουμε με ανησυχία την αξιολόγηση τη Κομισιόν για τα ωφέλη αυτών των συμφωνιών με τη Philip Morris International τις επόμενες εβδομάδες, όπως αναφέρατε κι εσείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε όμως ακόμη πιο μακριά. Είναι σημαντικό τώρα να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται διαπραγματεύσεις. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώνεται για τις συζητήσεις. Συνεχώς. Και όχι μόνο όταν τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να μας προσκαλείτε και εμάς στην τράπεζα των συζητήσεων ως παρατηρητές για να παρακολουθούμε αν θα ήταν καλό ε, να καταλάβουμε και εμείς τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να παραταθούν αυτές οι συμφωνίες και να πιστούμε ότι είναι καλό να παραταθούν αυτές οι συμφωνίες. Γιατί πρόκειται για λεφτά των φορολογουμένων. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αίσθηση στο κοινό ότι απλώς τους κρατάμε στην πάντα για κάτι το οποίο είναι τεράστιο, ε, τεράστιο διακύβευμα και οικονομικός και αλληλαίος πώς για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτως ή άλλως οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Και πώς θα εκπροσωπηθούν αν δεν ενημερώνεται και δεν συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Σωστά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, δύο λεπτά. Δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ την Επίτροπο για τη μεγάλη συνεδρίαση που έγινε και κλεισμένων των θυρών με συμμετοχή των, της Επιτροπής μας και για την ε, παρουσία της εδώ ε, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο των προϊόντων καπνού γιατί χάνουν και οι εθνικοί ε, προϋπολογισμοί και ο ε, Προπολογισμό της Ένωσης δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν ελέγχουμε δραστηριότητες πάση φύσεω και εγκληματική φύσεω, και που επηρεάζει την ε, υγεία όταν δεν ελέγχουμε τα όσα συμβαίνουν, μπαίνουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά, τα οποία είναι και πλαστά και στα πλαίσια αυτής της κρίσης δημιουργούνται καταστάσεις ε, ανεξέλεγκτης ανεξέλεγκτες που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες. Στις συμφωνίες θα πρέπει να έχουμε ε, συντονισμό για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτή, αυτό το λαθρεμπόριο. Για την ε, ομάδα μας, οι νέες συμφωνίες θα θέλαμε να γίνουν μετά από διαπραγματεύσεις ανοιχτές, αν προκύψουν συμφωνίες. Και θα, θέλαμε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν είναι χρήσιμε ή όχι, για να αποφύγουμε μεγαλύτερα δεινά. Θα πρέπει να έχουμε και έλεγχο και να δούμε και τι επίπτωση έχουν στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και την και τα πλαστά προϊόντα καπνού ε, και το λαθρεμπόριο. Και αυτό γίνεται βέβαια σε παγκόσμια κλίμακα. Ως ομάδα θα θέλαμε ε, βήμα-βήμα να παρακολουθούμε το διάλογο που κάνει η Κομισιόν, έτσι όπως απαιτείται από τη Συμφωνία. Και θα θέλαμε η γνώμη μας να ληφθεί υπόψη, ούτω ώστε να μην υπάρξουν μαξιμαλιστικές θέσεις που θα προκαλέσουν μεγαλύτερα δεινά. Δεν θα θέλαμε τέτοια τσιγάρα, ειδικά σε περίοδους ε, κρίσης θα θέλαμε λοιπόν αφού δούμε την έκθεση να επανέλθετε εδώ για να σας πούμε την γνώμη μας. Και ο βασικός στόχος των συμφωνιών θα πρέπει να είναι να προστατεύσουμε την υγεία, την φυσική υγεία, αλλά και την οικονομική υγεία ε, των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Ε, για λεπτά. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Το υποσυζήτηση θέμα είναι αμφιλεγόμενο και το ίδιο και ο σχετικός κανονισμός. Αφενός, δεν υπάρχει κανένα ε, γενικευμένο αίτημα για ανάπτυξη της βιομηχανίας. Το αντίθετο προσπαθούμε να περιορίσουμε τις δραστηριότητές της και προσπαθούμε να περιορίσουμε και τον αρνητικό αντίκτυπο επί της δημόσιας υγείας. Ε, ταυτόχρονα όμως είναι θεμητό να έχει δραστηριότητες αυτός ο κλάδος και άρα θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι όροι ανταγωνισμού και να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της αγοράς. Μην ξεχνάμε επίσης ότι προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό εισόδημα στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες να συναρμοστούν στα πλαίσια ενός κανονιστικού, ρυθμιστικού πλαισίου. Θα πρέπει να αλλάξουν κάποιες παράμετροι. Το θέμα της ε, δίκαιης ε, κατανομής των εισοδημάτων από τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις φαρμακοβιομηχανίες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Ε, συγγνώμη. Επίσης θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αυτές οι τρεις ε, συμφωνίες ε, είναι οι μοναδικές ε, που υπάρχουν και αν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα που υπάρχουν. Πώς θα έπρεπε να ενημερωθούμε καλύτερα για το περιεχόμενο τους και γιατί εκπνέουν διαφορετικές ημερομηνίες. Τρίτον, το λαθρεμπόριο ταξινομείται στην ίδια κατηγορία με άλλα φαινόμενα που δεν ρυθμίζονται όμως από αυτές τις συμφωνίες. Παραδείγματος χάρη κατακλυσμός της αγοράς με τσιγάρα χαμηλής ποιότητας, ε, τσιγάρα που πολλούνται εκτός της ρυθμισμένης αγοράς και προέρχονται από τρίτες χώρες. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Σόνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουγα με προσοχή την ε, παρέμβαση της συναδέλφου. Θα ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση. Όταν μιλάμε για αυτό τον αγώνα που γίνεται και το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα είναι τα λεφτά. Τα λεφτά και από πλευρά των κυβερνήσεων και από πλευρά αυτών που παραβιάζουν τον νόμο. Θεωρείτε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουν αναλυφθεί αρκετά μέτρα ούτως ώστε να παρεμποδιστούν τέτοιες δραστηριότητες στο μέλλον. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτησή σας. Ορθά υποδείξατε πως ε, η τρέχουσα πολιτική δεν επαρκεί. Ανέφερε ότι θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και αναφέρθηκα στην παρέμβασή μου μόνο σε τρία σημεία. Όμως αν είχαμε περισσότερο χρόνο μπορώ να σας μιλήσω και για άλλα. Για τη ρύθμιση της πολιτικής όντως θα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ευχαριστώ κύριο Ντεγιόγκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο για τις διευκρινήσεις και τη δήλωση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί το λαθεμπόριο. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Στην αρχή η συνεργασία με τις καπνοβιομηχανίες ε, ήταν ε, σε επίπεδο νομικής συμφωνίας και διευθετήσεων. Σήμερα έχουμε ε, φαινόμενα λόμπι, έχουμε την οδηγία τη σχετική για τα προϊόντα καπνού και τι βλέπουμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πάρα πολύ φιλικά παλικάρια, για να το πω έτσι. Δεν είναι τίποτα ευχάριστοι οι άνθρωποι. Και δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως συνηθισμένους λομπίστες ή κανονικές εταιρείες. Εγώ έχω κανόνες όταν έρχεται κάποιος από το λόμπι της καπνόβιομηχανίας στο γραφείο μου, θα πρέπει να το δηλώνω. Όχι μόνο ποιος είναι, αλλά και τι υλικό μου έχει φέρει, τι ε, συζητήσαμε. Ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είστε υποχρεωμένοι να μας διαβιβάζετε όλο το υλικό. Όχι μόνο σε εμά τους βουλευτές, αλλά και στην κοινή γνώμη, ε, στο λαό, οτιδήποτε σας διαβιβάζει η καπνοβιομηχανία. Και θέλω οπωσδήποτε να φτάνει στα χέρια των πολιτών αυτό το υλικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάς για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε οι συμφωνίες με τη Φίλιπ Μόρις θεωρήθηκαν σημαντικό στοιχείο στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Παρά τη συμφωνία και πολλές άλλες που ακολούθησαν με το Japan, το Tobacco, ε, ε, ε, British American και Imperial Tobacco Limited που είναι κολοσσή, χρειάζεται πολλής ε, χρόνος για να ακτιθούν αυτά τα διαφυγόντα κέρδη 10 δις που είναι από έσοδα από ειδικού φόρους κατανάλωσης κτλ. Αυτά τα ακούω χρόνια ολόκληρα. Ξέρετε ότι αυξάνονται οι επικρίσεις στο Κοινοβούλιο για τη συμφωνία αυτή. Ξέρετε την υπόθεση Ντάλι που συνδέεται με αυτό και την Μισελ Πετίτ που ήταν υπάλληλο ε, υψηλόβαθμος και έγινε σύμβουλος σε ένα δικηγορικό γραφείο που εργάζεται για τις εταιρείε αυτές ε, και τα θέματα τα σχετικά με την οδηγία δεν είναι ξένα προς όλα αυτά. Χρειαζόμαστε διαφάνεια. Όλα τα έγγραφα που έχετε για τις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να μας διαβιβάζονται. Είπε ο κύριος Σάβαρμα ε, με ποιο τρόπο είχαμε την ευκαιρία να τα δούμε και για πόση ώρα. Εγώ δεν αμφισβητώ τις συμφωνίες να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ε, με την ε, ε, τη Φίλιπ Μόρις, αλλά ε, εμείς συζητάμε και διαπραγματευόμαστε και εκείνοι προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σωστό και σύμφωνα με το άρθρο 5.3 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας θα πρέπει να ε, κοινοποιούνται όλα αυτά. Είναι χρήσιμες αυτές οι συμφωνίες. έχετε εξαγγείλει μια αξιολόγηση. Περιμένουμε πολύ μεγάλη περιέργεια και ενδιαφέρον να τη δω. Και όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ο Πρόεδρος διακόπτει. Ο κύριος Τσάνι έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν ξέρουν ότι τα κράτη-μέλη έλαβαν τα τελευταία δέκα χρόνια 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τι καπνοβιομηχανίε για να καταπολεμήσουν το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Δεν ξέρουν επίση ότι ένα μεγάλο βήμα των λαθρέων τσιγάρων προέρχεται απευθεία από τι εταιρείε που παράγουν προϊόντα καπνού. Και δεν ξέρουν ότι το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενεργοποιήσει διάφορε ε, ενέργειες, για κάνει διάφορες ενέργειες ε, κατά της Φίλιπ Μόρις που εγκαταλήφθηκαν το 2004 όταν μέσα σε 12 χρόνια αποφάσισε να δώσει ε, ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην Ευρώπη. Δεν ξέρουν επίσης πώς τα κράτη-μέλη εξόδεψαν αυτά τα κράτη-μέλη. Αυτό που ξέρουμε καλά είναι ότι ο καπνός από τα τσιγάρα είναι η δεύτερη αιτία ε, θανάτου στον κόσμο και η βασική αιτία ε, θανάτου θα μπορούσε να έχει αποτευθεί. 80.000 ε, άτομα στην Ιταλία ε, πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον καπνό. Ε, αν ήμασταν πονηροί θα σκεφτόμασταν ότι τα κράτη-μέλη και οι Κομισιόν δέχονται λεφτά από τις καπνοβιομηχανίες για να τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να πουλάνε καπνό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερόν για ένα λεφτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, για το λαθρεμπόριο έχω να πω ότι αυτό προέρχεται απορρέει άμεσα από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γενικευμένο λαθρεμπόριο καθίσταται δυνατό από το Σέγγεν με την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων. Ε, το Σέγγεν οδηγεί σε έκρηξη του λαθρεμπορίου προϊόντων του καπνού. Εσείς ευθύνεστε άμεσα για αυτό το φαινόμενο. Ε, Σέγγεν 1, Σέγγεν 2 ε, όπως εφαρμόζεται και στη Γαλλία με τον Σαρκοζή. Εγώ σας λέω ότι για να σταματήσει το λαθρεμπόριο πρέπει να καταργήσουμε το Σέγγεν, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο κάνουν. Όλα πρέπει να καταργηθούν. Ε, έχετε μία μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Από τον κύριο Σφάμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε Φερά, μετά από αυτά που αναφέρατε για το Σέγγεν, γνωρίζετε ότι το λαθρεμπόριο έχει να κάνει με την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, ενώ το Σέγγεν έχει να κάνει με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Μήπως τα έχετε μπερδέψει λίγο στο μυαλό σας. Αγαπητέ συνάδελφοι, όχι καθόλου δεν μπερδεύτηκα. Εγώ θεωρώ ότι όσο δεν έχουμε μια αποτελεσματική εσωτερική πολιτική, δηλαδή να αναλάβουν την ασφάλεια και τις, αστυνομικέ ε, αστυνομικές τους δυνάμεις ε, τα κράτη-μέλη, ποτέ δεν πρέπει να αναχαιτήσουμε το λαθρεμπόριο. Ε, Έχετε κι άλλη μπλε κάρτα. Από τον κύριο Λαβριγιού. Δέχεστε. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερθήκατε στο Σέγγεν και μόλις σας διευκρίνησε ο συνάδελφος Σουάμπ ότι δεν, προ... δεν εμπίπτει αυτό στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Σέγγεν. Υπάρχει και μια χώρα, η Αγγλία, που δεν είναι μέσα στο Σέγγεν. Εσείς δηλαδή ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει λαθρεμπόριο τσιγάρων στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου ε, μήπως ε, υπάρχει κάποια ανακολουθία σε αυτά που δηλώνετε. Απάντηση. Ε, κύριε Λαβρίγε, ας δούμε τι γίνεται στην ιστορία. Συγγνώμη, έχω ταργήσει όλα τα νομικά μέσα ελέγχου ε, κατά του λαθρεμπορίου, όχι μόνο των τσιγάρων. Δείτε και τι γίνεται με τους διακινητές στη Μεσόγειο. Εγώ πιστεύω ότι όσο δεν αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια νέα πολιτική για την ενίσχυση της κυριαρχίας των κρατών, δεν θα βγάλουμε άκρη. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γκρέσλε, δύο λεπτά. Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση είναι μια φυγή προς τα εμπρός και χαίρομαι πάρα πολύ που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτέλους δημοσίως ε, ε τοποθετείται μετά από δύο-τρία χρόνια αυτής της μυστικοπάθειας που τη διακατήχε. Και τώρα θέλουμε να δούμε τι απέφερε η συμφωνία. Έχουμε μειώσει το λαθρεμπόριο, στα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτές οι συμφωνίες δεν είναι συμφωνίες κατά πολέμησης απάτης και τίθεται το ερώτημα τι ακριβώς είναι. Είδαμε κάποια έγγραφα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, ε, με μεγάλα ελλείμματα ε, στην αλυσίδα ε, διανομής και σε καμία περίπτωση δεν είναι προστατευμένα από την απάτη. Και η Όλαφ έχει πιέσει ε, για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Με πραγματικά αξιοθαύμαστη υπομονή και επιμονή και για μας το σημαντικότερο ε, πρόβλημα είναι ότι η Όλαφ και οι αρμόδιες αρχές δεν βρίσκονται επί τόπου, δηλαδή στο Καλίνιγκρατ ή στην Κίνα. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Υπάρχουν προβλήματα παντού στον κόσμο. Ε, θα πρέπει να δημοσιεύονται ε, όλα τα έγγραφα που δεν έχουν να κάνουν με εμπορικό απόρριτο ή βιομηχανικό απόρριτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούμε να αξιολογούμε τι είναι αυτές οι συμφωνίες. Και οι ε, θεμητές προσδοκίες των καπνοβιομηχανιών για τις ετήσια επιπλέον πρόστιμα με βάση τις κατασχέσεις. Εδώ δεν έχουν να κάνουν αυτά τα θέματα με εμπορικό απόρριτο, εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω πουθενά. Ε, μετά, η συμφωνία. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα αν έχει τη θέση της η καπνοβιομηχανία στη Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Και ότι φέρουμε να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, δηλαδή είναι σε τέτοιο επίπεδο. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από την κυρία Γιάλα Σέντερ. Would Would you accept? Would you accept a blue card? Oh. Yes. You have the. Sí, sí, gracias, presidente. Sí, ευχαριστώ. Για να καταλάβω την επιχειρηματολογία του συναδέλφου, γιατί άλλο είναι η... το ότι κάνει ο Λάφα, ότι κατάσχει, ας πούμε, τσιγάρα και άλλα τι εμφανίζεται στα έγγραφα. Λοιπόν, θα ήθελα να σα ρωτήσω. Στη χώρα μου επικυρώσαμε το πρωτόκολλο για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού στα πλαίσια τη σύμβαση του ΠΟΗ για τον έλεγχο τη εργασία. Η κυβέρνησή σα όμω δεν το επικύρωσε. Γιατί η κυβέρνησή σα, κατά την άποψή σα, κυρία Γκλέσλε, δεν επικύρωσε αυτό το πρωτόκολλο. Δεν την ενδιαφέρει ή για άλλο λόγο. Το λέω για να καταλάβω καλύτερα. Για ποιου λόγου και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις, για να καταλάβω και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις συμφωνίες. Κοιτάξτε, απλούστατα. Εγώ δεν εκπροσωπώ την κυβέρνησή μου, είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είμαι εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βον για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ε, καλωσορίζω τις ε, συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών ε, της Κομισιόν και των τεσσάρων των μηχανιών για να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο στα προϊόντα καπνού και στο τσιγάρο. φυσικά υποφελούνται και οι καπνοβιομηχανίες φυσικά, γιατί χωρίς αυτές τις συμφωνίες αυτές οι εταιρείε θα έχαναν έσοδα. Φυσικά έχουν κίνητρο λοιπόν να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες. Αλλά είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να μειώσουμε ε, την απώλεια ε, εσόδων από τα, τους φόρους κατανάλωσης και γενικά τους ε, ειδικού φόρους. Ελπίζω λοιπόν οι συμφωνίες αυτές να συνεχιστούν και αυτές που θα εκνεύσουν σύντομα θα ανανεωθούν. Μην ξεχνάμε όμως τη διάσταση της υγείας και της ασφάλειας αυτών των συμφωνιών. Είναι σημαντικό να περιοριστούν τα, αυτού του είδους τα προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά για λόγους υγείας. Και βεβαίως θα πρέπει να σταματήσει ε, η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων από τέτοια προϊόντα, από το λαθεμπόριο τέτοιων προϊόντων, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εγώ υποστηρίζω ε, το να κάνει η Κομισιόν μία αξιολόγηση για... και, να μας... και να μας εξηγήσει, αν όχι τώρα, τον Ιούνιο ε, τις επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών. Ε, Επίση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπογράψουν το πρωτόκολλο για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο σε προϊόντα καπνού και τσιγάρα. Είναι σημαντικό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Όχι μόνο εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το παράνομο εμπόριο που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το εξωτερικό. Είναι σημαντικό λοιπόν για αυτό το λόγο να επικυρωθεί το συγκεκριμένο πρωτόκολλο από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Έχετε μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γκίλ. Ευχαριστώ κύριε Βόν. Δέχεστε ότι οι καταναλωτές της Ουαλίας εξυπηρετούνται καλύτερα από ανοιχτά σύνορα που επιτρέπει ε, την εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα καπνού. Ε, φυσικά, εάν κλείσουν τα σύνορα, ε, ή μάλλον αν είναι ανοιχτά τα σύνορα, ε, είναι πολύ πιο εύκολο να μπουν τα προϊόντα αυτά. Φυσικά δεν έχουμε σύνορα φυσικά γιατί είμαστε νησί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι τμήμα του Σέγγεν, όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, και εγώ ξέρω και εσείς ξέρετε, επειδή ταξιδεύουμε συχνά, ότι υπάρχουν, ότι ρούνται οι κανόνες ε, με αυστηρό τρόπο στα σύνορα. Είναι πολύ δύσκολο να περάσει λαθρέα οτιδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς μιλάμε για συμφωνίες με τις καμπτοβιομηχανίε, ώστε να γίνει ακόμα πιο δύσκολο στο μέλλον και, στην Ευρω... και για αυτούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για αυτούς που είναι εκτός να φέρουν αυτά τα παράνομα αγαθά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ρη, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, μπορούμε μετά από 12 χρόνια εμπειρία να αποτιμήσουμε και τη συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρις το 2004. Βλέπουμε ότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των όσων θέλαμε. Βλέπουμε ότι επιδιώκεται μείωση του λαθρεμπορίου, όμως από αυτά που διαβάζω και ακούω από τους εμπειροχνόμενες μας λένε τα αντίθετα. Ακριβώς το 2012 4 εκατομμύρια έδωσαν οι μεγάλοι 0, κάτι από την, το συνολικό όγκο πωλήσεων ε, ε, παραποιημένων τσιγάρων και μας λένε όλοι ότι νομίμως ε, όλα βαίνουν αισίως. Έτσι μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα έλεγα ότι τίποτα δεν βαίνει αισίως. Έχουμε και το άρθρο 5 για τη σύμβαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση σχέση ανάμεσα σε πολιτικούς ηθήνους και τους τέσσερις μεγάλους και με την κυρία Μακάβεν είχαμε ζητήσει να τηρηθεί κατά κατά γράμμα ε, η σχετική σύσταση. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να πω κλείνοντα ε, πώ έχουμε χρόνο να απορρίψουμε αυτή τη συμφωνία και να χρησιμοποιήσουμε ανταυτού τα πολύ αποτελεσματικά εργαλεία που ανέφερε η συγκήτρια. Σα ευχαριστούμε. Ο κ. Σαζολίκα θέλει να σα κάνει μια ερώτηση με τη διαδικασία τη μπλε κάρτα. Δέχεστε, όχι. Πολύ ωραία. Ο κ. Μποβέ, 1,5 λεπτό. Επίτροπε επανέρχομαι στη βασική αρχή, την πρώτη αρχή του πρωτοκόλλου του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Υπάρχει βασική σύγκρουση θεμελιώδου σημασίας ανάμεσα στα συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας και αυτών των αρχών που υπερασπίζονται τη δημόσια υγεία. Άρθρο 17, εδάφιο Γ της Ιδίας Σύμβασης, αναφέρει ξεκάθαρα ότι τα συμβαλόμενα μέρη, εκ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απορρίπτουν η αδίποτε εταιρική σχέση, η αδίποτε συμφωνία με τις καπνοβιομηχανίες. Ε, νομίζω ότι νομικός πώς ε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εάν συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, αντιβαίνουμε στο ευρωπαϊκό αλλά και στο διεθνές δίκαιο, στη Διεθνή Σύμβαση που προσυπογράψαμε το 2004 και η οποία ετέθησε ισχύ το 2005. Συντρέχει νομικός λόγος για να διακόψουμε τις διαπραγματεύσεις. Ας μη συγχαίουμε την απάτη με την παραποίηση. Η απάτη οργανώνεται από την καπνοβιομηχανία έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη από αυτά, ενώ με την παραποίηση χάνουν χρήματα. Και επειδή χάνουν χρήματα, στρέφονται προ τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπληρώσουν ε, τη χασούρα του. Δεν πρέπει να υποστηρίζουμε λοιπόν του απαταιώνε, ε, την καπνοβιομηχανία εννοώ, γιατί πρόκειται για πραγματική μαφία. Θα ήθελα ξεκάθαρα λοιπόν να απευθύνω σήμερα έκκληση. Διακόψτε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την καπνομηχανία διότι αντιβαίνει στο δημόσιο συμφέρον και στο διεθνές δίκαιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Ζανσολίκα θέλει να σας ε, υποβάλει μια ερώτηση. Δέχεστε. So this time he's... Πρόεδρε, νομίζω ότι ε, η κυρία Ρίς δεν θέλει να απαντήσει διότι δεν είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή της. Αυτό προκύπτει. Οπότε αυτού εγώ θα αντιθέσω στον κύριο Μποβέ την ερώτησή μου. Λοιπόν, ε, μας λέτε χρειάζεται διαφάνεια τεκμηρίωση. Ταυτόχρονα όμως δεν πιστεύετε πως οι αστυνομικέ δυνάμεις, οι Υπουργοί Εσωτερικών, τα τελωνία στα κράτη-μέλη πρέπει να μετέχουν σε αυτό το λαθρεμπόριο, διότι εγώ διάβασα ότι υπάρχει ανοχή από πλευρά του για το λαθρεμπόριο. Όμω πρέπει να κάνουν πρώτα απ' όλα δουλειά του να σταματήσουν να ε, συμμετέχουν σε αυτό. Απάντησα από τον κύριο Μπόβε. Συμφωνώ απολύτω. Θα πρέπει να επιτελέσουν το έργο του. Όμω ε, αυτά τα χρήματα που παίρνει η Όλαφ και τα ανακατανέμει στα κράτη-μέλη μέσω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα χρήματα που προκύπτουν από τη Συμφωνία των Κρατών μελών που ελέγχουν εξ ονόματος της ε, καπνοβιομηχανίας ε, τον έλεγχο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι μαφιόζοι ε, τον έλεγχο των παραποιημένων στην αγορά. Μα είναι σκάνδαλο αυτό. Δεν είναι ο ρόλος τους αυτός. Και βλέπουμε πως στα πλαίσια των δικαστικών αρχών, στο Βέλγιο συγκεκριμένα, στην υπόθεση Ντάλι, Βλέπετε τι έγινε, διακόπτει ο πρόεδρος τον κύριο Μπόβε. Κόμπορν, δύο λεπτά. Ε, thank you, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως θέλουμε να καταπολεμήσουμε ε, την ε, παραποίηση και το λαθρεμπόριο, αλλά όταν έχουμε ορθάνικτες τις θύρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πώς το καλό θα ελέγξουμε την ποιότητα και θα χαλιναγωγήσουμε το λαθρεμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βάζει το πιστόλι στον κρόταφο στις καπνοβιομηχανίες για να τις πληρώσουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Το ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο το λαθρεμπόριο, αλλά πώς προτείνετε εσείς να το αντιμετωπίσουμε για τα πλαστά ε, και τα παραποιημένα τσιγάρα ελέγχεται ε, το πακέτο των τσιγάρων. Αυτό θα ήταν το όνειρο του κάθε πλαστογράφου αν είναι ενιαίο ουδέτερο το πακέτο. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουν παραποίηση στα τσιγάρα. Ε, βγάζουμε τα περίπλοκα ε, ε των ε, ετικετών και των διαφόρων ε, δικτών ε, που βάζουν σε περίπλοκα πακέτα οι εταιρείε για να εξασφαλίσουν την ποιότητα. Όταν τα καταργήσετε όλα αυτά, πώς θα προστατεύετε τους καταναλωτές. Τσιγάρο θέλουν να καπνίσουν, καπνό και μόνο και όχι ποιο ξέρει τι βάζουν εκεί μέσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται σημαντικές συμφωνίες και λαμβάνει μεγάλα ποσά τα οποία ε, σπαταλάει με τελείως αντιδημοκρατικό τρόπο αντί να τα δίνει στα κράτη-μέλη. Τρεις συμφωνίες 2,15 ε, δισεκατομμύρια ευρώ έχουν συμφωνήσει να πληρώσουν οι εταιρείε. Αυτά είναι τύπου αλκαπόνε του Μακαρίτη μέθοδη. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα ρυθμίσει όλα αυτά. Thank you, Ευχαριστώ, κύριε Κόμπορν. Κυρία Κλαούντια Σμιτ, ένα λεπτό. Ähm, Ευχαριστώ. Ε, οι συμφωνίε ε, τώρα υποτίθεται ότι είναι καλές, λέτε κυρία Επίτροπε. Μπορεί να είναι στο χαρτί, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η συμφωνία με τη Φίλιπ Μόρις θα εκπνεύσει το 2016. Εξού και ρωτώ εγώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού βλέπει την προστιθέμενη αξία των ετησίων ε, πληρωμών ε, εάν ε, και εφόσον δεν είναι στοχευμένες αυτές οι πληρωμές και δεσμεύονται τα κράτη-μέλη που θα τα δαπανίσουν. Έχετε αρχίσει να συζητάτε με τη Φίλιπ Μόριτς για την παράταση συμφωνίας, αν όχι πότε. Και πότε θα κάνετε ένα ευρωβαρόμετρο που να ρωτάει ε, τους πολίτες πού είναι η προστιθέμενη αξία και τι άποψη έχουν για τα προϊόντα καπνού. Σορεύουν ε, τα ερωτήματα, συγκεντρώνονται και ο χρόνος τελειώνει. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκάιερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Αντιπρόεδρε Γεωργίευα, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Εγώ είμαι ένας χαρούμενος Γερμανός σοσιαλδημοκράτης. Και όταν τελειώσω την ομιλία μου θα έχετε καταλάβει τη διαφορά ε, μου από τον συνάδελφο Μποβέ. Ε, να πω κάτι που δεν ακούστηκε ακόμα. Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων είναι πολύ σημαντική διότι από πίσω κρύβονται δομές οργανωμένου εγκλήματος. Ε, θα πρέπει αυτό το υλικό να εισαχθεί, να διανεμηθεί. Τα χρήματα τα παίρνουν μετρητά. Θα πρέπει να τα ξεπλύνουν, να μπουν στην κανονική νόμιμη κυκλοφορία. Όπω γίνεται σήμερα το λαφρεμπόριο δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε ένα οργανωμένο έγκλημα. Και αυτό είναι κάτι που υπονομεύει ω κατάσταση τη δημοκρατία και ε, είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Είναι γεγονό ότι ο μεγαλύτερο κίνδυνο δεν είναι από τι μεγάλε εταιρείε ε, ε, στο μεταξύ κυκλοφορούν ε, φτηνά παράνομα τσιγάρα. Cheap whites είναι κάτι που δεν πουλιέται στη Γερμανία πουθενά νόμιμα και έχει φτάσει κατανάλωση στο 25% του συνολικού όγκου. Καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. λοιπόν, για να περιοριστεί το εμπόριο χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. Δεν αρκούν αυτές οι συμφωνίες. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίζει την Όλαφ και να στέλνει και συνδέσμους σε σημαντικές χώρες παραγωγούς όπου ήδη βρίσκονται βιομηχανίες και έχουν επαφή και με τις ε, κρατικές αρχές. Η Όλαφ εκπροσωπείται στην Ανατολική Ευρώπη τώρα μόνο στο Κίεβο. Δεν είναι δυνατό αυτό. Ε, λοιπόν, οι συμφωνίες έλεγα είναι ένα και μόνο μέτρο. Δεν συμφωνώ με τον συνάδελφο των πρασίνων ούτε με τους χριστιανοδημοκράτες που λέγουν ότι θα πρέπει να διακοπούν οι συνομιλίες σε καμία περίπτωση. Δεν, τι θα κάνουμε. Με εκκλήσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ε, τους πιέσουμε εκεί που τους πονάει, δηλαδή στην τσέπη τους. Έχετε γαλάζια κάρτα του κυρίου Μποβέτη, δέχεστε. Ναι. Μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Όταν μίλησα για τη διαφορά ανάμεσα στην απάτη και την παραποίηση, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγνωρίζει ότι η απάτη είναι οργανωμένη. Ας πούμε από την ίδια τη Φίλη Μόρις. Είναι σαφέστατο αυτό. Τα δίκτυα που υπάρχουν στην Ευρώπη από την ε, Ρωσία ας πούμε ε, στο παρελθόν και τώρα και από άλλους διάβλους αυτό είναι αναγνωρισμένο οι ίδιοι οργανώνουν την απάτη. Αυτό που είναι πρόβλημα σήμερα για αυτούς είναι η παραποίηση, γιατί χάνουν χρήματα με την παραποίηση, ενώ με την απάτη όχι. Το σκάνδαλο λοιπόν σήμερα είναι αυτό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά ανάμεσα στα δύο. Ενώ η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία αναγνωρίζει σαφέστατα την ευθύνη ε, της Φίλιπ Μόρις στο ίδιο το λαθρεμπόριο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μποβέ. Ο κύριος Γκάιερ. Βεβαίω και καταλαβαίνω τη διαφορά, αλλά αγαπητέ συνάδελφε, θα πρέπει και εσεί να παραδεχτείτε ότι στο μεταξύ ε, το ποσοστό των Φίλιπ Μόρι στις κατασχέσεις ε, έχουν μειωθεί κατά 85% τα τσιγάρα. Αυτά που λέτε λοιπόν για την κατάσταση και τα όσα λέγει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, είναι κάπως ξεπερασμένα, δεν είναι επίκαιρα στοιχεία, διότι η αιτίαση αυτή ότι οι ίδιοι υποστηρίζουν το λαθρεμπόριο, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν ισχύει το οργανών. Γι' αυτό σας ε, υποστηρίζουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Μύροσλαφ Ποχέ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, κάτι την άποψή μου το αν καπνίζει κάποιο ε, κάνει μεγάλο κακό στην υγεία του. Είναι από του μεγαλύτερου κινδύνου. Οτιδήποτε κάνουμε για να περιορίσουμε αυτόν τον κίνδυνο είναι ευπρόσδεκτο. Ε, Επίση, ε, κάτι άλλο τώρα για το παράνομο εμπόριο ε, προϊόντων καπνού. Προφανώ εκεί χάνονται εκατομμύρια ευρώ, αλλά υπάρχουν και άλλε αρνητικέ συνέπειες. Σε ορισμένα κράτη-μέλη το κάπνισμα ε, δημιουργεί φοβερή εξάρτηση ειδικά στους νέους. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι τα έσοδα από αυτό το ε, εμπόριο ε, οδηγούν στην άξιση του εγκλήματος. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και θα πρέπει να του δώσουμε μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλωσορίζει τις συμφωνίες που έγιναν το 2004. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια θετική προσέγγιση για τα, τα βήματα που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες που θα μας ενημερώσουν καλύτερα για το μέλλον αυτών των συμφωνιών. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, αν αυτές οι συμφωνίες ε, πέτυχαν αυτό που ελπίζαμε χρόνια πριν παρότι οι διαπραγματεύσεις με τις καπνοβιομηχανίες ε, ξεκίνησαν εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω, δεν έχουμε λάβει καθόλου πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποια θα είναι η κατάσταση ε, τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουμε ιδέα εάν η συνεργασία με τις καπνοβιομηχανίες είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου αυτή η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι θετική. Δεν μπορεί έτσι να πείσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος ε, Μπαλτζίτης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το 2007 στις συζητήσεις στην Ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτησε τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Φίλιπ Μόρις και τις συμφωνίες γενικά με άλλες ε, καπνοβιομηχανίες που θεωρήθηκαν επιτυχής. Έγιναν πολλά για να καταπολεμηθεί το παράνομο εμπόριο ε, τσιγάρου ε, και το λαθρεμπόριο σε σχέση με το 1990 χάνονται δισεκατομμύρια ε, ευρώ ετησίως και τα περισσότερα τσιγάρα ε, μπαίνουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση από το εξωτερικό και στη Βαλτική το ίδιο δημιουργείται έτσι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα σε αυτό το ε, τομέα. Για να πάρουμε θέση όμω, αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τι συμφωνίε αυτέ με τι καμπιτοβιομηχανίε μετά το 2016, όταν επνεύσουν οι τρέχουσε, θα πρέπει να ακούσουμε πληροφορίε για ό,τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα και ποιε ήταν οι ελλείψει των ε, τρεχούσων συμφωνιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλόρες. Ένα Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Εκπλήσω λίγο που ε, ε, λέτε ε, αυτούς τους ανθρώπους λαθρεμπόρους. Είναι εγκληματίες. 20 χρόνια τους ξέρω, ψηφίσαμε και την οδηγία και τώρα αρχίζουμε να χαλαρώνουμε τα κριτήρια ιχνηλασιμότητας και να δίνουμε στις εταιρείες ευκαιρίες για μεμονωμένες ε, συμβάσεις. Είναι λάθος. Θα πρέπει επιτέλους να κάνουμε αυτό που ζητήσαμε πριν από ένα χρόνο και αποφασίσαμε. Να έχουμε μια στρατηγική για την ιχνηλασιμότητα. Και θέλω να πω μερικά πράγματα. Η καπνοβιομηχανία, ιδιαίτερα αυτή που μιλήσατε προηγουμένως, αυτή, έχουν μεγάλο συμφέρον να συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα ανείχνευσης και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ δηλώνουν πολλά ε, λαθρέα και λίγα παραποιημένα. Γιατί ε, όπως είχε το σύστημα έπρεπε να πληρώνουν. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε πια στα παιδιά μας ότι υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα ε, σε αυτό τον αιώνα με συγχωροχάρτια. Και μην βιάζεστε πάρα πολύ να, ε, και μην επιταχύνετε να ε, παραταθεί η συμφωνία. Τα είπε και η κυρία Γκρέσλε, δεν θέλω να τα επαναλάβω, με κάλυψε τους ήταν πολύ καλά τα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτές οι συμφωνίες δεν είναι τέλειες και έχουν ε, γίνει αντικείμενο κριτικής ε, από πολλές πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο Κυρίω ε, για τη στενή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην καπνοβιομηχανία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε έχει υπάρξει και παρελκυστική πολιτική σε σχέση με την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας ε, για τα προϊόντα καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των παραποιημένων τσιγάρων και της παράλληλης αγοράς ε, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και από ουσία άλλων μέτρων θα έπρεπε νομίζω κατά τη γνώμη μου να καλωσορίσουμε με προσοχή ναι μένα αλλά να καλωσορίσουμε την παράταση αυτών των συμφωνιών. Φυσικά μπορούμε, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Θα πρέπει να ε, περιορίσουμε την ζήτηση ε, αρχικά. Αυτή την ιδιαστική συνήθεια θα πρέπει να την αποτρέψουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ούτως ώστε ε, ταχύτατα να εφαρμοστεί η οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στην ε, διαδικασία ε, Catch the Eye. Θα δώσω σε, το λόγο σε έναν αναπολιτική ομάδα μόνο, γιατί έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο. Η κυρία Πέτερ. Ευχαριστώ. Ε, συνιστούν ε, άμεσο κίνδυνο για την υγεία τα τσιγάρα και θα πρέπει ε, όχι μόνο να ελέγξουμε αυτά τα προϊόντα αλλά και το λαθρεμπόριο που συνδέονται και με απώλεια εισοδήματος σε επίπεδο εθνικού προϋπολογισμού. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για τα λεφτά των φορολογουμένων. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες και άρα οφείλουμε να έχουμε περισσότερη ενημέρωση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την καπνοβιομηχανία. Το λαθρεμπόριο είναι ένα συχνότατο ε, έγκλημα που διαπράτεται ε, στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται και με τη ε, φτώχεια που επικρατεί σε πολλές ε, τέτοιες περιοχές. Χρειάζεται στοχευμένη πολιτική. Ευχαριστούμε. Νέκοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Πάνω από δέκα δις ετησίως χάνονται εξαιτίας του λαθρεμπορίου. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας ε, πρωταρχικά για να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Πέραν αυτού παραβιάζονται συνθήκες εργασίας, ε, κανόνες της κοινωνικής νομοθεσίας ε, και ούτω καθεξής. Ε, στη Βουλγαρία παραδείγματο χάρη πάνω από 10 εκατομμύρια τόνοι τσιγάρων εισάγονται λαθρέα. Ε, πάνω από 150.000 χάνονται από τον 150 εκατομμύρια χάνονται από το φόρο ε, ειδική κατανάλωσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να εξυπηρετήσουμε άλλους κοινωνικούς στόχους. Διακόπτη ο πρόεδρος ε, Μπάσκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Κατακρίνουμε εκτενώς τις συμφωνίες με την καπνοβιομηχανία. Εξπακούεται ότι δεν είναι τέλειες, αλλά είναι απαραίτητες όπως και η σωστή εφαρμογή των συμφωνιών. Η Βουλγαρία είναι μεγάλος παραγωγός προϊόντων καπνού. Το 13% των εισοδημάτων στο γεωργικό τομείο προέρχονται από τον καπνό και στην απασχόληση το 5% απασχολείται σε αυτόν τον κλάδο και σε ορισμένες κοινότητες είναι μοναδική πηγή εισοδήματος. Όλα τα περιοριστικά μέτρα λοιπόν για την καπνοβιομηχανία θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο την αγορά της Βουλγαρίας για τα προϊόντα καπνού. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τον ελέγχο για τη σωστή εφαρμογή των συμφωνιών που στόχο έχουν την αναχέτηση του λαθρεμπορίου. Ευχαριστούμε. Γιάκοψιτς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι συμφωνίες θα θέσουν τέρμα στην παραποίηση και στην απάτη. Αν ναι, τότε είναι ευπρόσδεκτες. Εάν λύσουν το πρόβλημα απώλειας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τους εθνικούς προπολογισμού θα είναι ευπρόσδεκτες. Αλλά, Επίτροπε, όπως βλέπετε, υπάρχουν ε, υποψίες ότι δεν θα το καταφέρουμε τόσο εύκολα αυτό το πράγμα. Λόγω των εμπλεκόμενων σε όλη αυτή την ιστορία. Θα ήθελα να επωφεληθώ από αυτή την ευκαιρία που έχω και να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω να δώσετε προσοχή όχι μόνο στους μεγάλους ε, παραγωγούς καπνού και προϊόντων καπνού, αλλά να προστατεύσετε επίσης και τους πιο μικρούς. Γιατί αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ σημαντική, παραδείγματο χάρη για την περιοχή μου και τη χώρα μου. Στην Κροατία παράγουμε καπνό και τσιγάρα. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τους υπόλοιπους, όχι μόνο τους μεγάλους, στο πακέτο συμφωνιών. Ο κύριος Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Επίτροπε. Αναμφισβήτητα υπάρχουν διάφορες διαστάσεις που θα πρέπει να διευκρινίσει σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες που συνάπτεται με την ε, καπνοβιομηχανία. Υπάρχουν επίσης ε, πτυχές που πρέπει να διευκρινιστούν σε σχέση και με το περιεχόμενο, το αντικείμενο των συμφωνιών ε, για το λαθρεμπόριο των προϊόντων καπνού, διότι πρόκειται για τη βιομηχανία που προσδιορίζει αν είναι παραποιημένα ή όχι, γιατί όχι ένα εξωτερικό εργαστήριο, παραδείγματος χάρη ένα εξάρτητο εργαστήριο. Υπάρχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα με την καπνοβιομηχανία και πρέπει οπωσδήποτε να ε, δώσετε περαιτέρω διευκρινήσεις. Ε, επίσης, ε, ε, υπάρχουν, ε, τα, υπάρχει το θέμα των ποσών και της ανακατανομή τους στα κράτη-μέλη και εκεί χρειάζονται διευκρινήσεις. Ε, πολλά πρέπει να κάνουμε για την καταπολέμηση του φαινομένου. Παραδείγματο χάρη σε τέσσερα χρόνια στην Πορτογαλία, παραδείγματο χάρη μειώθηκε στο ίμιση ο αριθμός των μαγαζιών που μπορεί κάποιος να καπνίσει. Βλέπουμε ξεκάθαρα ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από όλη αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γεωργίευα, αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα σας ξεχωριστά και όλους μαζί για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη συζήτηση. φαίνεται ε, ξεκάθαρα πόσο περίπλοκο είναι το θέμα που απόψε συζητούμε. Θα ήθελα και πάλι να ζητήσω συγγνώμη για τη σύγχυση προσώπων και κομμάτων. Δεν ε, ήταν εσκεμμένη. Ευχαριστώ τον κύριο Στάς και τον κύριο Γκάιε για τα όσα είπαν. Θα ήθελα να σας πω τα εξής πέντε σημεία και να σας εξηγήσω σε ποια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε σε μια ε, διαρκή συζήτηση που έχουμε με το Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Έχω δεσμευτεί προσωπικά για να συνεργαστούμε από κοινού να δούμε ποιο ακριβώς είναι εκείνο το μέσο και εργαλείο που χρειαζόμαστε. Όπως πολλοί από σας είπατε, χρειαζόμαστε μια ευρύτερη προσέγγιση. Δεν εξαντλείται ούτε περιορίζεται στο συγκεκριμένο αυτό εργαλείο, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το ρόλο της για το μέλλον. Πρώτο ήταν αυτό. Δεύτερον, μπορεί να διήστανται οι απόψεις, αλλά ένα θέμα κυριάρχησε και βρίσκει τους πάντες σχεδόν σύμφωνους. Και αυτό είναι η ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια. Όσο λοιπόν προχωρούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα γίνεται μια ανοιχτή και δημόσια συζήτηση. Βέβαια, στο βαθμό που μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια σε αυτό το θέμα. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε θα προσπαθήσουμε να προτείνουμε τρόπους για να έχετε κι εσείς πιο ενεργό συμμετοχή στη διαδικασία αυτή. Τρίτον, δεν διεξάγονται αυτό τον καιρό διαπραγματεύσεις. Καμία όπως προβλέπεται από τη συμφωνία, είχαμε κάποιες διερευνητικές συνομιλίες για να βολιδοσκοπήσουμε τη Philip Morris International ε, δύο χρόνια πριν την εκπνοή της συμφωνίας ε, θα πρέπει ενδεχομένως να εξτάσουμε το θέμα της παράτασης. Αυτές οι διερευνητικές συνομιλίες ασχολήθηκαν με ένα αποκλειστικά θέμα εάν ε, εκφράζει ενδιαφέρον η Philip Morris να παραταθεί η συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρονται. Και εμείς είπαμε, ε, εκατέρωθεν δηλαδή και οι δύο πλευρές, ότι πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε βήματα υπέρ ή κατά των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να ε, ολοκληρώσουμε την αξιολόγησή μας, η οποία ε, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, είναι καθοδόν. Θα σας ενημερώσουμε λοιπόν βάσει της αξιολόγησης ανάλογα και σε διαβούλευση και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο αν θα προτείνουμε παράταση ή όχι. Κάποιες φωνές ακούστηκαν εδώ σαφώς υπέρ, ε, κάποιοι με μεγαλύτερη σαφήνεια, κάποιοι πιο επιφυλακτικά και προσεκτικά θεώρησαν ότι είναι χρήσιμο το εργαλείο και ακούστηκαν και φωνές ξεκάθαρα κατά. Θα πρέπει να εξετάσουμε το κόστος και το όφελος πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε απόφαση. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει με τρόπο διαφανή και δημόσιο. Δεν πρόκειται να υπάρξουν κρυφές διαπραγματεύσεις που δεν θα τις μάθετε εσείς. Σε περίπτωση που υπάρξουν καν, διότι και αυτό είναι ανοιχτό. Τέταρτον, μια ερώτηση που μου έγινε και θέλω να απαντήσω άμεσα αν έχουμε ερωτήσατε το δικαίωμα να σκεφτούμε καν τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο άρθρο 5.3 της Συμφωνίας Σύμβασης ε, καλεί τα μέρη να προστατεύουν τη δημόσια υγεία τους από εμπορικά ή άλλα συμφέροντα. Και μάλιστα κάποιος είπε να μην τους μιλάτε καν. Εσείς δεν το είπατε, να μην ε, συζητάτε μαζί τους. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η γραμματεία της έχουν εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς ε, θέλουν να εφαρμόζεται από τα συμβαλόμενα μέρη το ελόγο άρθρο και γίνεται ρητή ε, εξαίρεση για δεσμευτικές συμφωνίες όπως είναι αυτές οι περιπτώσεις προϊόντων καπνού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ε, αστόχαστα και επιπόλαια να προχωρήσουμε στη συμφωνία αλλά υπάρχει μια διευκρινιστική οδηγία Πέμπτο και τελευταίο θέμα. Και εδώ μια διευκρίνηση για το ανεξάρτητο εργαστήριο. Συμφωνήσαμε ότι είναι απαραίτητο, το αναφέρατε κάποιοι από εσά. Δηλαδή δεν μπορούν οι ίδιες εταιρείε να είναι και κριτές και κρινόμενοι για να κάνουν όλους τους ελέγχους. Και τότε είμαστε κάπως τυφλοί εμείς. Και σας επιβεβαιώνω ότι λάβαμε μια απόφαση να υπάρξει ένα ανεξάρτητο εργαστήριο που, στο οποίο θα μπορούμε να απευθυνόμαστε. Επίκειται λοιπόν η αξιολόγηση και θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι ήταν εντυπωσιακός ο αντίκτυπος στη μείωση του λαθρεμπορίου. Για να σας δώσω μια αίσθηση, ε, είχαμε εδώ μια συζήτηση μια μισή ώρα σχεδόν για αυτό το θέμα. Και κάθε λεπτό που συζητούσαμε ε, κατάσχονται 22 ε, παράνομα ε, πακέτα και ε, πρόκειται για όγκους δισεκατομμυρίων. Αυτά λοιπόν είναι πακέτα που δεν κυκλοφορούν στην αγορά μας κάτω της ε, νόμιμης τιμής. Είναι προϊόντα που δεν φτάνουν στα χέρια των νέων μας και ε, που δεν στερούν έσοδα από τους δημόσιους κορβανάδες. Είναι σαφέστατα τα ωφέλη, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι μεταβαλλόμενο και το τονίζω. Τώρα έχουμε αυτή την οδηγία και το πρωτόκολλο. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και συμφωνώ πολύ με εκείνους που το είπαν για να εφαρμοστεί η οδηγία. Να επιταχυνθεί η κύρωση του πρωτοκόλλου, και αυτό είναι και παραμένει ο μεγαλύτερος στόχος μας. Και το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουμε είναι στο ορατό μέλλον. Χρειάζονται και άλλα επιπλέον εργαλεία για να έρθουν να συμπληρώσουν τα δύο αυτά μεγάλα ε, θεμέλια που βάλαμε στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. για λόγους υγείας ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα και το λαθρεμπόριο για λόγους και υγείας και ασφαλείας και για φορολογικούς λόγους εσόδων. Και αυτό θα το κάνουμε με τη δική σας βοήθεια για την οποία σας ευγνωμονώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση.